Ε, Ο ψηφιακός κόσμος δίνει τεράστιες ευκαιρίες και για αναψυχή και για εργασία. Στη χώρα μου, ε, στη πόλη μου βλέπω ότι αναπτύσσονται ε, ψηφιακές ικανότητες ε, και βελτιώνει τη συνδεσιμότητα. Εξαιρετικές ευκαιρίες. Για να γίνει αυτό χρειάζεται υψηλής ταχύτητας ε, βριζονικό δίκτυο. όταν εργάζεται κανείς από το σπίτι βεβαίως μειώνονται οι αποστάσεις, τα μεταφορικά, όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Ε, υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία, όπως λένε οι ψυχολόγοι, ψυχολογικές επιπτώσεις. Να τις δούμε και αυτές. Στα πλαίσια των συστάσεων του ΟΣΑ, ταξινόμηση εργασίας κλπ. Και πολύ σημαντικό και είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στην Ευρώπη τώρα υπάρχουν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας νες, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Λεϊτάο Μαρκές. Ευχαριστώ πολύ. Το 1834 στο... Ε, ε, το 1934 πέρασαν ε, νόμοι ε, οι οποίοι ε, διασφάλιζαν την εργασία. Από τότε προχωρήσαμε πολύ. Φτάσαμε στην ψηφιακή εποχή που είναι μια μορφή βιομηχανικής επανάστασης. Η στροφή αυτή, η μετάβαση θα πρέπει να γίνει πιο γρήγορα και θα πρέπει να γίνει χωρίς αναταράξεις. Χρειάζονται περισσότερες δεξιότητες στις κοινωνίες θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ε, όλες τις κοινωνικές συνιστώσεις. Δεν πρόκειται μόνο για τα εργοστάσια, τις μονάδες παραγωγής, πρόκειται για την κοινωνική ζωή, την εργασία αλλά και προσωπικές σχέσεις. Κανείς δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με τρόπο δημοκρατικό και όλοι, όλα ε, θα πρέπει να ε, λειτουργούν με σύστημα δίκαιο. Χρειάζεται συνεργασία λοιπόν μεταξύ κοινωνικής πολιτικής και ψηφιακής οικονομίας. Ε, θα, πρέπει δηλαδή να παίξουμε συντονισμένα όπως ένα κονσέρτο του Μότσαρτ για πιάνο. Ο κύριος Στάγκα, ένα λεπτό. Γινόμαστε μάρτυρε μια ιστορική συγκυρία. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει τέσσερι ψηφιακέ στρατηγικέ την επόμενη εβδομάδα και με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί και η ψηφιακή αντεπα... αντεπανάσταση γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει τεχνητή νομοσύνη στο μέλλον. Έχουν το δικαίωμα επιχειρήσεις να εισβάλλουν στην ιδιωτική μας ζωή ή ε, θα πάρουν θεραλέα απόφαση να σκοτώσουμε αυτό το θηρίο. στην, στην το Google χρησιμοποιείται κατά 80% στα δημοτικά σχολεία. Επιθυμούμε να καθορίζει το Google τι μαθαίνουν τα παιδιά μας ή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για να μάθουμε τι μαθαίνουν τα παιδιά μας, εμείς ίδιοι. Ε, το ζητούμενο είναι η πρόθεση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής ε, στην ψηφιακή εποχή. Ας ε, δούμε τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον Επίτροπο κύριο Σμιτ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, άκουσα Τι συζητήσεις σας και διαπιστώνω ότι υπάρχει μια πλατιά συνένεση μεταξύ σας και για την ανάγκη να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την ψηφιακή οικονομία. Γιατί δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση για την Ευρώπη. Καμία άλλη εναλλακτική. Από την άλλη όμως να δώσουμε και τεράστια σημασία στις διάφορες πτυχές και στους διαφόρους κινδύνους που επιφέρει αυτού του είδους η οικονομία, αυτή η νέα οικονομία. Κοινωνική κίνδυνη, κίνδυνη σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, κίνδυνη κάποιες επιχειρήσεις να ελέγχουν τα δεδομένα. Δεν θα γίνουν όμως αυτά μοιραία. Μπορούμε να προωθήσουμε την ψηφιακή οικονομία και παράλληλα να υπάρξει κοινωνική προστασία, να υπάρξουν δικαιώματα, να υπάρξει προστασία των δεδομένων. Δεν θα πρέπει απλώς να υποστούμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Θα πρέπει να τη διαμορφώσουμε με βάση τις ανάγκες μας. Αφού άκουσα τις συζητήσεις σας, απευθύνεται μία πρόσκληση προς την Κομισιόν να δουλέψει πάνω στις δύο αυτές πτυχές, πάνω στους δύο αυτούς άξονες και θα παρουσιάσουμε αυτό το ψηφιακό θεματολόγιο όντω και παράλληλα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες για την προστασία και την εγγύηση των δικαιωμάτων. Προανήγγυλα ότι η Κομισιόν θα κάνει μια μεγάλη διάσκεψη για την εργασία στις πλατφόρμες και ελπίζω το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει. Είμαι πεπισμένος μάλιστα θα, θα συμμετάσχει, τόσο ώστε το ευρωπαϊκό μοντέλο σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Ήδη έχουμε δώσει παραδείγματα, έχουμε προστατεύσει τα δεδομένα. Θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε πάλι παράδειγμα με την κοινωνική προστασία, με τα κοινωνικά δικαιώματα προωθώντας αυτή την οικονομία, αλλά να την καθυποτάξουμε στην υπηρεσία του συνόλου. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Η κυρία Μπρντζάκ. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, η αρχή της ισότητας στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, οι δίκαιες εργασιακές σχέσεις, οι συνθήκες εργασίας αποτέλεσαν πολλές φορές το αντικείμενο νομοθεσίας, ψηφισμάτων κλπ. Είμαι βέβαιη ότι είμαστε στη σωστή πορεία. Αυτό που λείπει είναι ειδικέ στρατηγικές αφιερωμένες στην ψηφιακή ανάπτυξη. Αντιλαμβάνομαι από την Κομισιόν ότι αυτές οι προτάσεις σύντομα θα δοθούν. Περιμένω τις προτάσεις της Κομισιόν και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε γόνιμη και καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κλείνει η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η δήλωση της Επιτροπής για τη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων. Είναι δυνατόν να έχουμε catch the eye και μπλε κάρτες ε, με το ηλεκτρονικό σύστημα. Ε, υπάρχουν οδηγίες στην είσοδο της ε, Ολομέλειας. ήθελα... θα ήθελα να δώσω το λόγο κατευθείαν στην Κομισιόν. Ε, Επίτροπε Ντάλη, έχετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ που τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων την θέσατε στη σημερινή μερίσια διάταξη. Τους πρώτους μήνες μετά την ε, εντολή της Κομισιόν μπόρεσα να συναντήσω ήδη πολλούς από εσάς. Όλες οι αλλαγές, ε, όλες οι συναντήσεις επιβεβαίωσαν ότι όλοι μας είχαμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε αυτή την πολιτική. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που μου δείξατε ε, και δείξατε και στην Επιτροπή ήδη πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της χρειάζονται την πλήρη υποστήριξή σας ώστε να γίνει ε, ένας χώρος ισότητας η Ευρώπη ε, για τα φύλλα. Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης αρχή μας και η Ευρώπη είναι καλός, καλός, καλό μέρος για να ζει κανείς. Αλλά θα ήταν... Ε, υπερβολικό να πούμε ότι φτάσαμε εκεί που θέλουμε, γιατί υπάρχει ακόμα μισθολογικό χάσμα. Μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρώπη έπεσε θύμα ε, σεξουαλικής ή άλλης βίας από την ηλικία των 15 και αυτό αφορά εκατομμύρια γυναικών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις αποτρόπες ανισότητες η πρόεδρος Βαντερ Λάιεν, η αρμόδια επίτροπος, ε, είμαστε ε, δεσμευμένοι υπέρ της πολιτικής ε, για την ισότητα. Και η στρατηγική για την ισότητα των φύλων είναι ένα ακόμα βήμα. Αρχές Μαρτίου θα γίνει δεκτή θα υπάρξουν πολιτικές δεσμεύσεις, θα υποστηριχθούν στρατηγικά, ε, συστηματικά έργα για την ισότητα στην ε, Ευρώπη ε, και ευρύτερα. Έχουμε φιλόδοξη στρατηγική και το πλαίσιο μιας κίνηση ορατήσε που αντιτάσσεται στα δικαιώματα των γυναικών που υπάρχει στην Ευρώπη και διεθνώς τα τελευταία χρόνια ε, θα πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να τονίσουμε την συνεχιζόμενη δέσμευσή μας, τη δέσμευση της Κομισιόν υπέρ της ισότητας των φύλων. Έγινε ευρεία διαβούλευση για τη στρατηγική και δημόσια διαβούλευση που πήρε, δέχτηκε πάνω από 1.300 απαντήσεις. Η ισότητα των φύλων είναι οριζόντιο θέμα. Η στρατηγική θα, θα ε, προωθήσει την δυτή μας στρατηγική, ε, συνδυασμένη δηλαδή με στοχευμένες δράσεις σε επιμέρους θέματα. Θέλουμε μια πιο συστηματική προσέγγιση στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού της πολιτικής για να εντάξουμε την ε, διάσταση του, της ισότητας σε όλες τις πολιτικές. Επί της ουσίας θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα όραμα προσανατολισμένο προς το μέλλον για μια Ευρώπη ε, με ισότητα, όπου οι άνδρες και οι γυναίκες, τα γόρια και τα κορίτσια με όλες τις διαφορές τους θα είναι ελεύθεροι από βία και στερεότυπα με βάση το φύλλο. Θα έχουν την ευκαιρία να ευημερήσουν στην αγορά εργασίας, να τεθούν επικεφαλής ε, της πολιτικής, των επιχειρήσεων και να συμμετέχουν ισότιμα σε όλους τους τομείς. Σημαντικές οριζόντιες ε, σκέψεις που θα υπογραμμιστούν στη στρατηγική είναι να αμφισβητήσουμε τα στερεότυπα ε, που υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά τα θέμα, η στρατηγική θα τονίσει τις προτεραιότητες ε, που υπάρχουν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, οικονομική ενίσχυση των γυναικών, μείωση του μισθολογικού χάσματος, μέτρα υποχρεωτικά, δεσμευτικά, ε, ανάδειξή του σε διοικητικά συμβούλια, αναγνώριση του έργου ε, των, γυναικών που εργάζονται στο σπίτι, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ε, επίσης θα πρέπει να προσυπογράψουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και καθυστερεί παρά τις προσπάθειές μας. Θα υποβάλλουμε νομοθετικές προτάσεις για να ενισχύσουμε την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων και να καταπολεμήσουμε ε, κάθε μορφής ε, ε, βία κατά των γυναικών. Θα πρέπει να ενταχθεί στον κατάλογο των αξιόπινων πράξεων στην ψηφιοποίηση επίσης ε, και στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να εντάξουμε τα θέματα αυτά. Μαζί με την ε, υιοθέτηση της πολιτικής συνδέουμε ε, μια διαδικασία διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς για δεσμευτικά μέτρα διαφανή που θα υποβάλλουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Γνωρίζω ότι εισάγοντας ε, αυτά τα μέτρα διαφάνειας, αυτό μπορεί να αποτελεί πρόκληση και πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία για τέτοιες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των εργοδοτών, των εργαζομένων και των εθνικών διοικήσεων. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας και να συζητήσω μαζί σας. Ελπίζω πραγματικά να τύχω της υποστήριξής σας, ούτως ώστε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε αυτό το άλμα που χρειάζεται τόσο πολύ προς μια Ευρώπη ισότητας των φίλων στην εργασία και στην ε, ζωή. Ευχαριστούμε τώρα εκ μέρου του ΕΛΚΑ για 1,5 λεπτό η κυρία Φράνσεν παρακαλώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο της Επιτροπής ε, για το γεγονό ότι η ισότητα των φίλων συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα αυτό είναι μία από τι θεμελιακέ αξίε ε, επί των οποίων δράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 67,4% δείχνει ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε. Θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Τα ταλέντα των γυναικών συχνά παραμένουν αναξιοποίητα και μια περικτική στρατηγική των φύλων περιλαμβάνει τρία σημεία. Δημιουργία ευκαιριών για τις γυναίκες, ε, ένταξη των γυναικών σε ένα ραγδαία μεταλλασσόμενο κόσμο, ψηφιοποίηση, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή κλπ. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες πλατφόρμες, νέες μεθόδους εργασίας. Ε, επίσης θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου την πιο δύναμη θέση των γυναικών και να ε, στηριχθούμε στη στρατηγική των ε, φίλων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να κλείσουμε το συνταξιοδοτικό και μισθολογικό χάσμα. Θα πρέπει να συμπελάβουμε τις γυναίκες στις επιχειρήσεις να ε, ξεπεράσουμε πλεονεκτήματα που βασίζονται στο φύλλο και να αποκτήσουμε και να φροντίσουμε για μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή, ούτω ώστε οι γυναίκε να πάρουν τι ευκαιρίε που του ε, αξίζουν, ούτω ώστε όλα, η έκφραση είναι θετική για όλου. Εκ μέρου των σοσιαλιστών ε, η κυρία Νότσιλ, ευχαριστώ πολύ. με κυρία Πίτροπε, μας έχετε στο πλευρό σας. Εάν ε, πρόκειται για ουσιαστικές ε, πρόοδους στην εξίσωση των φύλων, θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να, να πω ότι οι γυναίκε δεν είναι αδύναμε, αλλά αποδυναμώνονται βάσει παραδόσεων και στερεοτύπων. Δεν είμαστε αδύναμε. Η αποδυνάμωση έρχεται απ' έξω. Εάν δούμε τώρα τη στρατική, η οποία όπω ε, ε, ε, ελπίζουμε θα δερθεί στην Ευρώπη έχουμε τα εξή αιτήματα. Θέλουμε μια αυτοδύναμη στρατηγική, με ένα ξεκάθαρο στρατηγικό σχέδιο. Θέλουμε να δούμε ε, ξεκάθαρα βήματα. Δεν θέλουμε οπισθοδρομήσει και δεν θέλουμε να παραβιάσουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Θέλουμε την ίση μεταχειρίση των φύλων και την, τον τερματισμό όλων των μορφών διάκριση. Επίση, όπω το τόνισε η Επίτροπο, ε, επιθυμούμε να γίνει κάτι τέτοιο σε όλου του πολιτικού τομεί. Ε, στη φορολογική πολιτική, την ψηφιακή πολιτική, την ε, κλιματική πολιτική, τον προπολογισμό, την έρευνα, τη γεωργία κλπ. κλπ. Ε, η ισότητα των φύλων αφορά όλους τους τομείς της πολιτικής και θέλουμε να δωρεθεί ταυτόχρονα σε όλους. Δεν θα αναφερθώ στην πρόληψη ε, των αγώνα κατά της ε, βίας έναντι των γυναικών ή τη συμβατότητα μεταξύ επαγγελματική και προσωπικής ζωής ή τα σεξουαλικά δικαιώματα. Θα ήθελα να θέσω το επίκεντρο της ομιλίας με ένα άλλο θέμα τη διασύνδεση μεταξύ ίσης μεταχείρισης των φύλων και δημοκρατίες. Και εδώ, κυρία Επίτροπε, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ζητούμε, ζητάμε να υπάρξει μια μελέτη η οποία οποία να αναλύσει τις εθνικιστικές πολιτικές στη βάση της ισότητας των φύλων. Και ζητούμε τα δικαιώματα των γυναικών να αναλύονται σε όλες, σε όλες τις χώρες μέλη και να υπάρξουν οι αντίστοιχε εκθέσεις. Η ισότητα των φύλων συναρτάται με, την, το κράτος δικαίου. Και εκεί όπου παραβιάζεται, παραβιάζονται και οι κανόνες του κράτους δικαίου. Ευχαριστούμε εκ μέρους του Ρινιού για δύο λεπτά η κυρία Τολερέ, παρακαλώ. Ε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τη δεσμευσή σας, για την εργητικότητά σας, για να τελεσφορήσει αυτή η στρατηγική υπέρ της ισότητας. Ήταν πραγματικά η κατάλληλη στιγμή. Έχει τεράστιες προκλήσεις μπροστά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε όμω για να προωθήσει οτιδήποτε να γίνει πραγματικότητα η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ισότητα στην υγεία. Το 1974 ε, νομιμοποιήθηκαν οι αμβλώ στη χώρα μου. Όμω το 2020 υπάρχουν ακόμα άνδρε και γυναίκε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν ίση και δωρεάν πρόσβαση στην άμβλωση και δεν έχουν και εκπαιδευτική και εκπαίδευση για θέματα σεξουαλικά διότι το θέμα της υγείας αυτό είναι πολύ σημαντικό και όλοι θα πρέπει να είναι ίσοι στο θέμα της υγείας. Η αναπαραγωγική και η σεξουαλική υγεία όταν παραβιάζεται, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα γεμότα των γυναικών και αυτό θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε αμήλικτα. Ας μιλήσουμε για αυτές τις παραβιάσεις, θα πρέπει να τις εκριζώσουμε, να ξεκινήσουμε από τις οικονομικές παραβιάσεις. Χθες μιλούσαμε για τις γυναίκες επιστήμονες και ερευνητές. Όμως υπάρχει τρομερή ε, μισθολογική διαφορά μεταξύ άνδρων και γυναικών σε, στη δουλειά. Και η διαφορά αυτή είναι πολύ πιο έντονη στη σύνταξη. Θέλουμε ίση εργασία και τότε ίσο μισθό. Οποιασδήποτε και αν είναι οι προελεύσεις, οι πεπιθήσεις καν, καθενός, θα πρέπει όταν οι γυναίκες να, όταν κάνουν την ίδια δουλειά να παίρνουν τα ίδια λεφτά. Επίσης δεν θα πρέπει το γεγονός ότι οι γυναίκε τεκνοποιούν να τιμωρούνται γι' αυτό. Θα πρέπει να μην τιμωρούνται. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα στην καριέρα, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε θέσει εξουσία. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να δώσει απτά φρούτα, αυτά αποτελέσματα και έχουμε παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όταν υπάρχει ισότητα δεν θίγεται σε τίποτα οι επιδόσεις των ε, επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε τη φυσική βία. Μπλοκάρεται η σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης γιατί υπάρχουν απροθυμίες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει το Συμβούλιο να δώσει απαντήσεις ε, για να σταματήσουν διάφορες μορφές βίας. Θα πρέπει να έχει μία προσέγγιση αδέκαστη και τελειώνοντας θέλω να σας πω με το σύμφωνο Σιμών Βέι ξεκινήσαμε από τις ισχύουσες νομοθεσίες της ε, χώρας Ένωσης ε, να διδαχθούμε από τις χώρες που έχουν εξασφαλίσει την ισότητα για να την ε, εξασφαλίσουμε και στις υπόλοιπες χώρες παντού σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Να σας θυμίσω ότι πρέπει να τηρείτε τον χρόνο. Κριστίνα Άντερσον τώρα. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι βάσει βάση των κανονισμών ε, απαγορεύονται σύμβολα και σημαίες. Λοιπόν, ε, αφαιρέστε παρακαλώ τη σημαία, απευθύνομαι στην συνάδελφο που θα λάβει το λόγο και θα πρέπει να υπενθυμίζετε και από τους ε, υπαλλήλους, ότι αυτό απαγορεύεται. Λαμβάνω υπόψη ότι φοβάται πάρα πολύ τις εθνικές ε, σημαίες στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ντροπή ε, να πρέπει να απομακρυνθεί η σημαία. Μιλάμε πάντως για την στρατηγική ισότητας. Υπάρχει ισότητα ε, όλοι ε, γεννόμεθα με τον ίδιο τρόπο, οι γυναίκες και οι άνδρες, αυτό δεν αμφισβητείται. Αν και άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια αξία, έχουν διαφορετικές τάσεις, ε, αδυναμίες και δυνατά σημεία. Είναι διαφορετικές οι προκλήσεις. Οι άνδρες θα, ε, ε, έχουν και εκείνοι ε, τα προβλήματά τους. Γιατί δεν ενθαρρύνει η Κομισιόν την, τους άνδρες να είναι άνδρες και τις γυναίκες γυναίκες. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα ισότητας από τα κράτη-μέλη. Όχι, θα πρέπει να υπαγορεύεται κεντρικά. Η, οι, οι, οι οικογένειες θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα φέρνει τα λεφτά στο σπίτι, ποιος θα ασχολείται με τα παιδιά η, η, Κομισιόν στο τέλος ε, θα ε, ε, εκπονήσει νομοθετική πράξη για το θυλασμό που θα πρέπει να γίνεται σε δίκαιη βάση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης, δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν αποφάσει των γυναικών να παραμείνουν στο σπίτι και να ασχοληθούν με την οικογένειά τους. Η θα πρέπει να ε, δούμε το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στα φορτηγά ή σε καθαρά ε, τομείς που κυριαρχούνται από τους άνδρες. Ας σταματήσουμε να θέλουμε να επανεκπαιδεύσουμε ε, σε βασικά θέματα τους άνδρες και τις γυναίκες. Αφήστε τους ανθρώπους να είναι άνθρωποι ξανά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που βγάλατε και τη σημαία. Δεν φοβόμαστε τίποτα, αλλά είναι κανονισμοί που ισχύουν για όλους. Η κυρία Κούνκε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλά μπορεί κανείς να πει για αυτό το θέμα, μακρύς ο κατάλογος. Ε, ως ε, πράσινη πολιτικός ε, βλέπω μια έλλειψη που είναι σημαντική δεδομένων των προκλήσεων, των μεγάλων προκλήσεων του κλίματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από τις αλλαγές στο κλίμα λόγω των ε, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Για να μπορούμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά τη Συμφωνία του Παρισιού χρειάζεται ε, ισότητα. Η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν όταν έγινε πρόεδρος είπε ότι την ισότητα θα την έβαζε με κεφαλαία γράμματα στη, στο θεματολόγιο και παρουσίασε και την Πράσινη Συμφωνία. Ε, δεν ανεφέρθηκε όμως στην ισότητα στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας. Και η αρμόδια επίτροπος για την ισότητα, η Ελένα Ντάλη, δεν ήταν παρούσα κατά τη συζήτηση αυτή. Γι' αυτό εγώ και η πράσινη ομάδα ζητήσαμε δύο πράγματα από την Ελένα Ντάλη. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, θα πρέπει να προωθήσει την πράσινη συμφωνία η οποία πρέπει να εφαρμόζεται ξεκάθαρα. Πρέπει να πάρουμε θετικά σήματα, θετικές ενδείξεις και ε, ε, προσβλέπω σε καλή συνεργασία με την Επίτροπο Ντάλι. Ευχαριστώ. Από το ECR, από την ομάδα ECR, η κυρία Βυσνιεύσκα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η ισότητα είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να είναι φιλόδοξη και ρεαλιστική ταυτόχρονα. Τι μορφή θα έχει νέα αυτή η αρχή. Υπάρχουν νέες προκλήσεις για να αντιμετωπίσουμε. Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος, του συνταξιοδοτικού κενού, ε, θα ήθελα να ε, προτείνουμε νομικούς κανόνες που θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν τις γυναίκες που θέλουν να συνδυάσουν επαγγελματική και, επαγγελματική, ε, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βίας κατά των γυναικών συμπεριλαμβανομένης της βίας στον κυβερνοχώρο, την πορνογραφία και το εμπόριο ανθρώπων. Δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες απειλούνται ε, με ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων και άλλα προβλήματα. Η νέα στρατηγική μας δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ακολουθήσει τη δική του αρχή που σημαίνει ένωση στη διαφορετικότητα. Ευχαριστώ. Και τώρα ε, ο Γκουέντζιέλ, η κυρία Περέιρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η στρατηγική ισότητα θα πρέπει να περνάει μέσα από την καταπολέμηση της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα για να καταπολεμηθούν αυτά. Οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ίση αμοιβή, ίση σύνταξη, ίσες συνθήκες εργασίας οι αντίστοιχες υπηρεσίες ε, ε, πρόσβαση στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. η ε, γονική άδεια που θα πρέπει να καταβάλλεται με τρόπο ισότιμο. Ε, συνδυασμός επαγγελματικής οικογενειακής ζωής χρειάζονται αντίστοιχοι μηχανισμοί για όλα αυτά, δυνατότητες ε, για που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους στην οικογένεια και στον εργασιακό χώρο. Ευχαριστώ. Η Ιζαμπέλα Αντινόλφη έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Συνάδελφοι, σε αυτή την αίθουσα μιλάμε πολύ για την ισότητα των φίλων και τα δικαιώματα τη γυναίκα. Αλλά α πούμε τα πράγματα ειλικρινά. Α παραδεχτούμε ότι δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ας, μάλιστα, πρέπει να δεχτούμε ότι οι γυναίκε αποδυναμώνονται και ταπεινώνονται. Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση, δεν υπάρχει μισθολογική ισότητα και στην Ευρώπη, σε πολλέ χώρε, η πορνεία είναι νόμιμη. Και αντί να καταπολεμήσουμε αυτή την κοινωνική μάστιγα, αποστρέφουμε το βλέμμα. Στην Ευρώπη υπάρχει ακόμα σκλαβιά για πολλές γυναίκες. Τις θεωρούμε εμπορεύματα προς αγορά και πώληση. Στην Ευρώπη οι γυναίκες σκοτώνονται και παραμορφώνονται από τους άντρες. Μπορούμε να επιβάλλουμε κανόνες. Στην πραγματικότητα είναι απλώς μια παρηγοριά, μια ανακούφιση, γιατί βασίζονται κυρίως σε ε, κυρώσεις προς τους παραβάτες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως είναι να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές. Γι' αυτό στρέφουμε προς τις μητέρες. Διδάξετε το σεβασμό προς τους άλλους. Μάθετε στα παιδιά σας, τα αγόρια σας να γίνουν άντρε με αλφα κεφαλαίο και στα κορίτσια σας να μην εξαρτώνται από κανένα και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, την ελευθερία τους φυσική και ηθική. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Ρώσα Εσταρά Φεραγκούτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε τη στρατηγική 2016-2019 για την ισότητα των φύλων. Ε, είχαμε. Και τώρα έχουμε τη νέα στρατηγική, η οποία θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα για αυτό το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να προχωρήσουμε με αποφασιστικό τρόπο. Ε, ούτως ώστε να πετύχουμε την ισότητα. Πρόκειται για ένα δημοκρατικό ζήτημα. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς ισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία ευημερία χωρίς σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ισότητα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα ε, να στηρίξουμε την ε, οδηγία της ε, εμφυλίωσης. υπάρχουν τρόποι να πετύχουμε αυτή την ουσιαστική ισότητα. Υπάρχει, επίσης υπάρχει και ένα θέμα ισότητα στη λήψη αποφάσεων, άρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία να είναι περιεκτικά, και προστά σε όλους. Επίσης, η βία κατά των γυναικών, οι τελευταίες στατιστικές μας λένε ότι δύο μεταξύ τριών γυναικών έχουν πέσει θύματα βίας. Υπάρχουν επίσης ζητήματα άλλα ε, τεχνητής ε, ε, ε παρενόχληση, συγγνώμη. Ε, έχουμε... Νομίζω ότι με τρόπο αυτό θα πετύχουμε να σταθούμε στο ύψος των ευρωπαϊκών αξιών. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για την δραστήρια στάση σας. Σας ευχαριστώ που προσπαθείτε να παρουσιάσετε το συντομότερο δυνατόν τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων και σας εύχομαι καλή τύχη με αυτή τη στρατηγική. Όμως, πρέπει να εκφράσουμε μια σαφή θέση για το τι πρέπει να περιλαμβάνει η στρατηγική. Καταρχάς, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για να καταπολεμήσουμε τη βία εναντίον των γυναικών και να εφαρμόσουμε την ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των γυναικών. Στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία αποπειραθήκαμε να συντονίσουμε και να συμφιλιώσουμε την ε, ιδιωτική και την επαγγελματική σφαίρα. Και καλούμε τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στην εσωτερική του νομοθεσία σωστά τη σχετική οδηγία. Επίση, το μισθολογικό και το συνταξιδοτικό χάσμα θα πρέπει να κλείσει. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε συγκεκριμένε αποφάσει. Η ευχή που σα εκφράζω είναι να τα καταφέρετε για να γίνει πραγματικότητα αυτή η στρατηγική. Η κυρία ο κύριος Ροντρίγκες Ράμος, για ένα λεπτό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στρατηγική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και σήμερα περισσότερο από ποτέ γιατί αναδύονται ολοκληρωτικές ιδεολογίες στην Ευρώπη ε, που αρχίζουν να επιτίθενται στα δικαιώματα και στις ελευθερίες των γυναικών. Το χειρότερο φαινόμενο βεβαίως είναι η βία. Και η χειρότερη μορφή βίας κατά των γυναικών είναι οι δολοφονίες, οι δολοφονίε γυναικών που αυξάνονται στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να είμαστε ε, ξεκάθαρη. Έχουμε ε, τελματώσει στην ε, συνθήκη της Κισταντινούπολης και πρέπει να υπογραφεί περισσότερες χώρες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη στρατηγική, κυρίως όσον αφορά δύο θεμελιώδη στοιχεία. Το ένα είναι τα δεδομένα. Κυρία Επίτροπε, δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει στη διάθεσή της δεδομένα, να γνωρίζουμε τους αριθμούς της πραγματικότητας της άσκησης βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη. Έχουμε περιορισμένα δεδομένα ε, και βάσει του άρθρου 11 της Συνθήκης Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να, ξεκινήσουμε, να προχωρήσουμε για να έχουμε δεδομένα συγκρίσιμα, για να ξέρουμε ακριβώς ε, ποια είναι ε, η πραγματικότητα του φαινομένου της βίας. Θα πρέπει να δώσουμε ένα όνομα, να την ονοματίσουμε. Ε, ένα κακούργημα, έγκλημα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένη ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο και ε, το Κοινοβούλιο είναι τέρος σας στον δρόμο αυτό. Ευχαριστώ. κυρία Λίτση, μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Κύριε Πίτροπε, στηρίζουμε τη σημασία της ισότητας των φύλων. Είναι κοινή μα αξίας. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, ας προσπαθήσουμε για να την προωθήσουμε σε όλες τις πολιτικές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κάνουμε την πολιτιστική επανάσταση, όχι σαν μία επιβολή. Τα φράγματα στη δουλειά εναντίον της γυναίκας ε, πλήττουν ε, την ανάπτυξη. Θα πρέπει να αρθούν οι φραγμοί. Το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη δείχνει ότι η ισότητα των φύλων θα προωθεί στην οικονομική ανάπτυξη. Όμως το Ινστιτούτο ε, αποτιμά σε αριθμούς, σε ποσά την ε, συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Ε, αν συμμετείχαν οι γυναίκε, ε, θα είχαμε 10 ε, εκατομμύρια περισσότερου εργαζόμενου στην αγορά Το θέμα είναι τι ισορροπία θα έχουμε στι οικογένειε. Η ισότητα των φύλων θα πρέπει να προωθηθεί και στι νέε πολιτικέ. στην ενιαία αγορά, στην ψηφιακή αγορά, στην τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί είναι πιο δραματικό το χάσμα. Θα πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο που διαχειρίζεστε τις πολιτικές. Γιατί και το ελεγκτικό συνέδριο θα εξετάσει την ένταξη της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δημοσιεύτηκε σήμερα η έκθεση που θα δημοσιευθεί την άνοιξη του 2021 για να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν οι πολιτικές Φοντερ Λάιν στον κόσμο των γυναικών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φουρτασούν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πέτροπε. Είναι σημαντικό ότι τελικά έχουμε μια στρατηγική. Κάποιος είπε προηγουμένω ότι η τελευταία στρατηγική τερματίστηκε το 2019. Ελπίζω έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία στρατηγική στη τελευταία θητεία. Και τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα έχουμε μια στρατηγική και ελπίζω να, είναι ένα, μια, να δώσει μια φεμινιστική όθηση. Κάτι που αναμένουν και οι Ευρωπαίοι πολίτε. Θα ήθελα να σα απευθύνω μια έκκληση να είναι φιλόδοξη σε διάφορου τομεί στο κοινωνιο-οικονομικό τομέα. Έχουμε την, πολλές ελπίδες με την υγεία περί διαφάνειας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με το, σχετικά με το θέμα της βίας. Η στασιμότητα όσον αφορά τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντινούπολης είναι απαράδεκτη. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο mainstreaming όλων των ε, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, γιατί θέλουμε το αποτύπωμα της ότας των φίλων παντού. Άρα, κυρία Πίτρο, παρακαλώ να κάνετε εσείς την διαφορά. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, η κυρία Μολντανόφσκα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Καλά νέα που ετοιμάζεται αυτή τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση πια. Μιλάμε για τεχνολογική πρόοδο, ψηφιοποίηση, αλλά ακόμα δεν έχουμε ισότητα σε ένα σημαντικό τομέα, όπως είναι τα φύλλα. Δεν υπάρχει ισότητα των φύλων. Το 2020 όλες οι χώρες θα έπρεπε να καταργήσουν τις διακρίσεις λόγω φύλου. Αν το κάναν αυτό, το ΑΕΠ θα αύξανε κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε διακρίσει βάρων των γυναικών. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και να το ανεχτούμε κοινωνικά και οικονομικά. Δεν μιλάμε μόνο για το μισθολογικό χάσμα. Δεν μιλάμε μόνο για τη φτώχεια που ε, προκαλεί. Ε, γιατί ε, το μισθολογικό χάσμα είναι μόνο 6%, ενώ στη σύνταξη η διαφορά είναι 35%. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις καριέρα όταν είσαι γυναίκα. Επομένως, η φτώχεια δεν μπορεί να έχει το πρόσωπο μιας γυναίκας πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίλβια Μόντικ. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πολλά θέματα θα μπορούσα να αναφέρω. Ε, εστιάζω όμως στη σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία σεξουαλική υγεία, η οποία είναι ένα δικαίωμα όλων των γυναικών ε, και των κοριτσιών, ανεξάρτητα από φιλή και ε, λοιπά. Αυτό πρέπει να εντάσσεται στην στρατηγική μας. Ε, επίσης, η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ένα άλλο θέμα είναι ποιος είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα των παιδιών. Ε, έχει αντίχτυπο αυτό στην ποιότητα της υγείας και της φροντίδας και τη φροντίδα επίσης των ηλικιωμένων. Υπάρχει ένα καινούριο σύστημα που έχουμε εισαγάγει εμείς, το οποίο προβλέπει ε, ποσοστώσεις ε, ε, και αυτό επηρεάζει και τη σύνταξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κομίν ή Ολιβέρες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι γυναίκε πάντα έκαναν διπλό αγώνα. Πάντα κουβαλούσαν δύο βάρη. Και το προσωπικό και το κοινωνικό. Οι γυναίκε είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Και παρόλα αυτά, ίσως και γι' αυτό υπάρχουν πολλές γυναίκες στην Ευρώπη που δεν έχουν εξασφαλισμένα τα δικαιώματά τους με αποτελεσματικό τρόπο. Τα τελευταία τρία χρόνια Κομισιόν, η διαφορά στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι στο 11%. 78% απασχόληση ε, στους άντρες, 66% στις γυναίκες. Υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στους μισθούς των ανδρών και γυναικών κατά 16%. Για να μην μιλήσουμε για, τις, ε, για τη βία κατά των γυναικών. Θέλουν μια κοινωνική αλλαγή οι γυναίκες για να εξασφαλιστούν απόλυτα τα δικαιώματά τους. Και αυτό μας αφορά όλους, και τους άνδρες και τις γυναίκες. Αν οι άνδρες δεν αλλάξουν το ρόλο που παίζουν στο δημόσιο βίο, στην επιχείρηση, στην οικογένεια, θα είναι αδύνατον οι οικογένειες, οι γυναίκες να απελευθερωθούν και να σταματήσει η παραβίαση των δικαιωμάτων τους και στις οικογένειες. Και το λέω από προσωπική εμπειρία. Ο φεμινισμός δεν είναι θέμα και υπόθεση των γυναικών, είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λουκατσιεύσκα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ντροπή που στον 21ο αιώνα οι Ευρωπαίες γυναίκες και οι γυναίκες όλων τον κόσμο μαστίζονται από τόσες ανισότητες. Γι' αυτό χαίρομαι, Επίτροπε, που είναι μία από τις προτεραιότητες της ε, τωρινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες των γυναικών από διαφόρους τομείς. Από την Ήπεθρο, τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες γιατί δεν μπορούν να βρουν θέση στα νηπιαγωγεία για τα παιδιά τους, ε, δυσκολίες ε, πρόσβασης στην υγεία, τις ηλικιωμένες γυναίκες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα στα γυρατιά τους. Υπάρχουν γυναίκες επίσης που δεν έχουν πρόσβαση σε, βασικά, σε βασικές θεραπείες για την υγεία τους. υπάρχουν γυναίκε που θέλουν να έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Και συχνά οι γυναίκες παρότι έχουν καλύτερη εκπαίδευση δεν βρίσκουν καλύτερη δουλειά ή δεν πληρώνονται το ίδιο με τον άντρα για την ίδια δουλειά όμως. Σκέφτομαι επίσης εκείνες τις γυναίκες οι οποίες πέφτουν θύματα μίσους, σεξουαλικής βίας, οικογενειακής βίας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προκλήσεις, γιατί δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Σκέφτομαι εκείνες τις γυναίκες που έχουν αναπηρία, που πρέπει να αντιμετωπίσουν φράγματα στην καθημερινή του ζωή. Εμείς ως Ευρωπαίες γυναίκες στο Ευρωκοινοβούλιο, παρά τις διαφορές μας, μπορούμε να μιλήσουμε με νέα φωνή για αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό για τόσες γυναίκες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο τον έχει ο κύριος Μάτιτς. Για ένα λεπτό. Και να σας υπενθυμίσω ακόμα μια φορά να σέβεστε το χρόνο που σας έχει δοθεί. Γιατί αλλιώς τον κλέβετε από κάποιον άλλον. Τον κλέβετε από αυτούς που έχουν ζητήσει ε, μπλε κάρτα ή συμμετέχουν στο Catch Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οι ευρωβουλευτές χαίρονται γιατί αυτή η στρατηγική δείχνει σαφώς τις νέες προτεραιότητες της Κομισιόν. Ζούμε σε εποχές όπου χρειάζεται να κάνουμε ε, βήματα ε, προς την αποφυγή της οπισθοδρόμησης στα δικαιώματα των γυναικών. Τα σεξουαλικά αναπαραγωγικά δικαιώματα ε, είναι εκείνα τα οποία πάσχουν περισσότερο. Υπάρχει επίσης και βία βάσει φύλου νομοθετικές διακρίσεις, έλλειψη εκπαίδευσης και όλα αυτά στηρίζονται σε πατριαρχικές αξίες που αντιβαίνουν στις δημοκρατίες μας. Αυτό που περιμένω από τη νέα στρατηγική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ότι δεν θα σταματήσει να είναι την πρώτη γραμμή για την ε, μάχη υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να μας γυρίσει πίσω στο μεσαίωνα. Αυτό είναι μια λιδία λίθος για μας. Κάτλιν Τσεκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται με βάση αυτή τη στρατηγική. Είναι πολύ σημαντικό. Να υπογραμμίσω ένα στοιχείο ε, τη βία κατά των γυναικών. Όταν μιλάμε για βία, συνήθως μιλάμε για αριθμούς. Μια στις τρεις Ευρωπαίες γυναίκες. Εγώ θέλω να μιλήσω για ανθρώπους. Εδώ έχουμε το πρόσωπο μιας ε, πολύ γενναίας γυναίκας η οποία ε, έπεσε θύμα βίαιης συμπεριφοράς από τον πρώην σύντροφό της. Ε, έπρεπε να τύχει νοσηλευτικής περίθαλψης, πολιτικής υποστήριξης και ε, λέμε πολλές φορές ε, ότι η προσχώρηση στη σύμβαση είναι, ε, δεν χρειάζεται. όμως βλέπουμε εδώ παραδείγματα γενναίων γυναικών που δίνουν τη μάχη τους και πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο. Και η Κομισιόν θα πρέπει να προσθέσει στον κατάλογο των αξιόπινων πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη τη βία, σωματική βία κατά των γυναικών και να προσχωρήσει η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Έχουμε κάποιους κανόνες εδώ στο Κοινοβούλιο. Μην τους ξεχνάτε. Δεν θέλω να χρησιμοποιείτε πόσταρ και αφήσει στο χώρο της Ολομέλειας, στις επόμενες παρεμβάσεις σας, γιατί οι κανονισμοί μας αφορούν όλους, ισχύουν για όλους. Και τώρα, το λόγο έχει η κυρία Ράιντκε. Όχι, ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρο. Η κυρία Τζιτζιμέντη. Έχει το λόγο. Για ένα μισή λεπτό. Η γυναίκα είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα τεράστιο έργο. Για την, λόγω της αποστολής της, λόγω της α, προσφοράς της υπέρ της ζωής και της ανθρωπότητας, για την καθημερινή της συμφορά, ε, συνεισφορά, με ευαισθησία, με γενεοδορία προς την οικογένεια και προς την κοινωνία και για την ε, δημιουργία μιας κουλτούρας που συνδυάζει την λογική με το συνέστημα. Χαρακτηριστικά της γυναικείας φύσης. Με αυτόν τον τρόπο η γυναίκα εμπλουτίζει την κατανόησή μας για τον κόσμο και συνεισφέρει σε μια αυθεντική διάσταση στις ανθρώπινες σχέσεις. Επίσης δίνει άοκνες μάχες για να υπάρχει ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά φράγματα που δεν επιτρέπουν την πλήρη υλοποίηση της ε, ισότητας. Η πραγματική γυναικεία χειραφέτηση είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το παραπέμψουμε πλέον στις καλένδες. Για όλες εκείνες τις γυναίκες που σιωπηρά ε, θυσιάζονται και δουλεύουν και ελπίζουν ότι θα ζήσουν ε, κάποτε την ισότητα και παρόλα αυτά ζουν μια εχθρική πραγματικότητα χωρίς δικαιοσύνη, με ταπεινώσεις και συχνά ε, δεν προστατεύονται στις ε, κοινωνίες ούτε καν η ζωή τους. Οι γυναίκες σιωπούν, ζουν τις ε, πίκρες αυτές μόνες. Γι' αυτό λοιπόν Είμαστε υπέρ αυτή τη πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων, που θα πρέπει να έχει δεσμεύσει ξεκάθαρε, ε, δείκτε ξεκάθαρου και ένα μηχανισμό παρακολούθηση, ούτω ώστε. Και διακόπτεται η ομιλήτρια από την Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ράιντκε. Για ένα λεπτό. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, στην πραγματικότητα είναι ένα μακρύ κατάλογο που θα ήθελα να συμπεριλάβω στο πλαίσιο αυτή τη στρατηγική ισότητα, αλλά θα εστιάσω την προσοχή μου σε δύο βασικά στοιχεία. Να, πρώτον, να υπάρξει ε, μια νομοθετική πρόταση όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα. Ε, χρειάστηκαν 63 χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, προκειμένου να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρόταση για την μισθολογική ισότητα. Δεύτερο θέμα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια οδηγία κατά της ε, βίας ε, απέναντι στις γυναίκες. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση με τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Μπολσονάρο η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα, προβλήματα, τα ιστορικά προβλήματα που έχουμε, όλα αυτά είναι πραγματικά ένα λίκνο ελπίδες, ελπίδας για, τους, για όλους τους μενιστές στον κόσμο. Και η στρατηγική αυτή είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ε, προσδοκίες που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα η κυρία Στέγκρουτ για ένα Fru talman! Jag är oerhört tacksam över tidigare generationers kvinnokamp och... πρόεδρε. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλα όσα έγιναν για τις γυναίκες. Σήμερα βλέπουμε ήδη τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Υπάρχουν όλο και περισσότερες γυναίκες στα πανεπιστήμια, στα ΜΜΕ κλπ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι λυπηρό που δίνεται μια άλλη εικόνα ότι οι γυναίκες είναι θύματα και συχνά λέγεται ότι είναι η ευθύνη της μιας πατριαρχικής κοινωνίας. Αλλά ο κίνδυνος της νέας στρατηγικής είναι ότι έχει έναν εσφαλμένο προ... προσανατολισμό. Ε, βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά όχι να εκχωρηθούν λάθος προνόμια. Δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε μια παλιά ανισότητα με μια καινούργια ανισότητα. Ε, το δικαίωμα ψήφου βεβαίως να υπάρχει. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κουντουρά για ένα λεπτό. Ε, κυρία Επίτροπε, για να πετύχει η στρατηγική σας για την ισότητα των φύλων πρέπει πρωτίστως να φροντίσετε να δεσμευτούν τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης σε ένα νέο πλαίσιο με κατευθυντήριες γραμμές και υποχρεωτικά συγκεκριμένα μέτρα για την ισότητα των φύλων προτείνω δεσμευτική νομοθεσία και συγκεκριμένα να κυρωθεί και να εφαρμοστεί χωρίς περιορισμούς η σύμβαση της κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη για να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών για να καταπολεμηθεί το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων να καμφθούν τα εμπόδια για την έγκριση Τη σχετική οδηγία για την ίση εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις που έχει παγώσει στο συμβούλιο από το 2013 να πάρθουν μέτρα πρόληψης αποτελεσματικέ διαφανεί, εμπιστευτικέ διαδικασίες καταγγελιών και αυστηρές αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των δραστών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. τέλος να συμπεριλάβεται ξεχωριστό κεφάλαιο στη στρατηγική για τις γυναίκες για την υγεία ώστε να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα της υγείας. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη εδώ και χρόνια δίνουν μάχη για την ισότητα των φύλων. Αλλά μέχρι στιγμή τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολιτικέ όχι απλώ δεν ήταν επαρκεί για να ξεπεραστεί το οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ε, πλήγμα που υφίστανται οι γυναίκε λόγω των διακρίσεων. Ο λόγο είναι πολύ απλό. Γιατί ο παραγωγικό και οικονομικό κόσμο ποτέ δεν θέλησε να παρέμβει στην, στο χώρο εργασία, εκεί όπου έχουμε συστηματικέ διακρίσει, καθημερινέ διακρίσει. Και επομένω, είναι πολύ σημαντική για μα αυτή η στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Γιατί είναι καινοτόμα σε ό,τι αφορά τι μεγάλε αλλαγέ που γίνονται, όπω η βιομηχανική και ψηφιακή επανάσταση. Αν δεν τη διαχειριστούμε σωστά, θα, δεν τις διαχειριστούμε σωστά αυτές τις ε, επαναστάσεις, θα αυξηθούν οι διακρίσει μεταξύ των γυναικών. Θα πρέπει να έχουμε όλα τα, μέσα, ούτως ώστε να σταματήσουν διακρίσει ει βάρο των γυναικών και στο χώρο εργασίας και για να παραμείνουν οι γυναίκες στο χώρο εργασίας. Ως κοινωνία των πολιτών και ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουν και οι ψυχικές και φυσικές ε, εκδηλώσεις βίας εναντίον των γυναικών. Θα ε, πρέπει να έχουμε μια στρατηγική στο ύψος όλων αυτών των προκλήσεων και θα στηρίξουμε όλες αυτές τις μάχες που είναι θέμα πολιτισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Μαρία Walsh. Ένα λεπτό. Επίτροπε εντάλληλοι συνάδελφοι, χαιρετίζω τη στρατηγική για την ισότητα. Η προώθηση της ισότητας θα πρέπει να είναι βασική δράση της Ένωσης. Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης για τις κοινέ μας αξίες και στόχους. Καθώς εξελίσσεται η κοινωνία, είναι σημαντικό να εντάξουμε την αρχή της συνένεσης. Ε, η βία κατά των γυναικών και ο καταναγκασμός είναι προβλήματα που αντιμετωπίζονται με τοπικά. Πρέπει να στηρίξουμε τις γυναίκες και πρέπει να πιάσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, που είναι η εκπαίδευση, η κοινωνική ανάπτυξη. Ε, δεν θα πρέπει να εμποδίζονται οι γυναίκες στις αποφάσεις τους. Ε, είναι σημαντικό να έχουν ίση θέση στην κοινωνία για να έχουμε μια ανεκτική κοινωνία. Ευχαριστώ, Επίτροπε Ντάλη, που πήρατε την πρωτοβουλία και αναγνωρίζω και τη συμβολή των πολλών αρένων συναδέλφων που μας βοηθούν. Σας ευχαριστούμε. Αν δεν συνεργαστούμε θα πέσουμε σε ότα μη ακουόντων. Ευχαριστώ. Πίνα Πιτσέρνο, η επόμενη ομιλήτρια. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Με μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Τώρα, μάλιστα, άναψε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγες εβδομάδες θα έχει τη δική της στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Αυτό είναι καλές ειδήσει. Επιπλέον, θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικέ ειδήσει αν λάβουμε υπόψη ότι στην τελευταία νομοθετική θητεία δεν είχαμε μια τέτοια στρατηγική. Επομένω, έχουμε θετική στάση στηρίζουμε αυτή την στρατηγική, σα, στηρίζουμε επίτροπε, μα αρέσουν αυτέ οι ειδήσει, γιατί η Ευρώπη είναι εκείνη η μεριά του κόσμου που έχουν τα περισσότερα δικαιώματα και έχουν λιγότερα, λιγότερες παραβιάσεις στα δικαιώματά τους. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Έχουμε διαφορές στους μισθούς και στις συντάξεις, λένε οι στατηγικές. Επίσης, ε, οι γυναίκες οι οποίες είναι σε διευθυντικές θέσεις είναι ελάχιστες και αυτό είναι γελίο. Ε, επίσης, ε, βλέπουμε στις εφημερίδες, στα κοινωνικά μέσα, ε, τι μόμπινγκ υπάρχει, τι παρενόχληση, τι βία κατά των γυναικών, κατά των κοριτσιών. Και αυτή είναι μια αδιανόητη κατάσταση, ε, ανυπόφορη για τη ζωή μας και την ελευθερία μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δεσμευτικά μέτρα, όχι ένα κατάλογο καλών προθέσεων. Δεσμευτικά μέτρα. Θέλουμε μια οδηγία, Επίτροπε, κατά της βίας. Μια οδηγία η οποία θα έχει δεσμευτικά μέτρα για να αποφύγουμε αυτό το δράμα που οι αδερφές μας σκοτώνονται από δολοφόνους που έχουν όνομα και πόνιμο, ε, που είναι θύματα όμως και μιας ε, πατριαρχικής και αρχα, ε, αρχαϊκής κοινωνίας. Κόβει η πρόεδρος στην ομιλήτρια και τώρα ο κύριος Πισλάρου έχει το λόγο για ένα λεπτό. Επίτροπε, Είχα ετοιμάσει μία επίσημη ομιλία, αλλά θα την αφήσω κατά μέρο για να στείλω ένα μήνυμα πιο συναισθηματικά φορτισμένο. Πολλές γυναίκες θεωρούν ότι το πρόβλημα ε, της ισότητας είναι σημαντικό, αλλά δεν το ε, συμμερίζονται μερικές φορές αυτό οι άνδρες. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές... Ε, μορφές βίας. Ε, εγώ το βλέπω καθημερινά. Έχω τέσσερα κορίτσια και τα εκπαιδεύω καθημερινά, ούτω ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να υπάρχει